Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, εμείς οι πρόεδροι της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και Θεμελιωδών Ελευθεριών χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαστε εδώ για την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Είναι σημαντικό θέμα η προστασία των νομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση νομοθετήματος. Έχουμε δύο εισηγητές από τις δύο επιτροπές οι οποίοι ισοτήμως εργάζονται για το θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Ε, να σας αναφέρω ε, γλώσσες έχουμε. Η συνεδρίαση πρώτα απ' όλα είναι δημόσια και μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Οπότε περνάμε και στο τρίτο ε, θέμα, έγκριση των πρακτικών της 22ης Ιανουαρίου 2014. Υπάρχουν ε, ε, παρατηρήσεις, όχι, ωραία. Οπότε μπορούμε απευθείας, εφόσον πρώτα διαπιστώσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά, να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Αλλά καταρχάς να δώσω το λόγο και στο συνάδελφο από την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για να μας πει ε, και αυτό το εισαγωγικό του σχόλιο. Äh, Ο συνάδελφος Λόπες Αγγίλαρ δεν θέλει να κάνει εισαγωγική ε, παρουσίαση, θέλει να περάσουμε στην ουσία να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στην εισηγήτρια της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, την κυρία Γκρέσλε, για να μας κάνει ε, την παρουσίασή της. Ευχαριστώ, λέει κυρία Γκρέσλε. Ε, χαιρετώ και, τους, ε, και τον συνεισηγητή. Έχουμε 100 τροπολογίες και δικές μας τροπολογίες και ε, τροπολογίες από τους συναδέλφους των δύο επιτροπών. Χτες είχαμε μια πρώτη συνεδρία των ε, σκιωδών και διαπιστώσαμε ότι δεν είχε έρθει κανένα σκιώδης. Αυτό μάλλον σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που θα έπρεπε να συζητηθεί μαζί μας. Οι δύο εισηγητές θα προτείνουν μια συγκεκριμένη γραμμή η οποία βασίζεται στα βασικά σημεία της έκθεσης, δηλαδή αυτά που έχουμε στην έκθεση, δηλαδή να υπάρχουν ε, ελάχιστες κυρώσεις ε, ΦΠΑ και οι μέγιστες κυρώσεις. Αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουμε και τις τροπολογίες. Δεν θα αποδεχτούμε λοιπόν τροπολογίες οι οποίες αποκλίνουν από αυτές τις αρχές. Θέλουμε λοιπόν να συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ στην οδηγία αυτή. Θέλουμε ελάχιστες και μέγιστες πίνας. Επιπλέον ε, θα συμπεριλάβουμε μερικά συμπληρωματικά, λίγα συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον προσθέτουν κάτι στην οδηγία. Δεν δεχόμαστε το θέμα της διεύρυνσης και προς άλλους τομείς. γιατί είχαμε και τροπολογίες. Έχουν διανεμηθεί και όλες οι συμβαστικές τροπολογίες και τις έχουν διάθεσή σας. Ε, βεβαίως ε, θα είχαμε θελήσει να συζητήσουμε με κάποιους συναδέλφους ορισμένε τροπολογίες γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι τις καταλαβαίνουμε αλλά έχουμε βεβαίως ακόμη δυνατότητα διμερών επαφών. Αυτή λοιπόν είναι η βασική μας κατεύθυνση που θα την ακολουθήσουμε και για τις τροπολογίες. Και έτσι ακριβώς με βάση αυτές τις αρχές θα διαμορφωθεί και ο κατάλογος ψηφοφοριών. Θα πρέπει να συζητήσουμε και μαζί με τη συνάδελφο Βέμπερ για να καθορίσουμε αυτή την ε, λίστα ψηφοφοριών και να σας τη στείλουμε για να μας πείτε αν έχετε επιπλέον παρατηρήσεις. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν συμφωνούμε για την νομική βάση, για την οδηγία. Η Επιτροπή Ελέγχου θέλει την 325 και η άλλη, η άλλη επιτροπή θέλει το 383. Και για το θέμα του Eurojust υπάρχει μια διαφορά απόψεων. Αλλά αυτά είναι τα μόνα δύο σημεία για τα οποία υπάρχουν διαφορέ απόψεων. Για αυτά λοιπόν τα δύο θέματα δεν θα υπάρξει κοινή σύσταση για την ψηφοφορία. Για όλα τα άλλα ναι. Κάθε ομάδα λοιπόν και κάθε ομάδα εργασία θα πρέπει να αποφασίσει κατόπιν ε, την άποψή της. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και για την πραγματικά καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Αγκρέσλε Να δώσω το λόγο στον επικεφαλής τη Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ, λέει στα γερμανικά ο κύριος Αγγιλάρ. Καλημέρα στα αγγλικά. Η κυρία Γκρέσλε νομίζω το έθεσε σωστά ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Ήταν καρποφόρα η συνεργασία μεταξύ μας. Είμαστε εδώ να εξετάσουμε τις τροπολογίες για την έκθεση περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να εξάρω το πολύ καλό έργο της εισηγήτρια και την πολύ καλή συνεργασία των συνεισηγητών. Μετά από παρατεταμένες συζητήσεις μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση που αντανακλάται στο σχέδιο έκθεσης. Δεν θα σταθούμε τώρα σε κάθε τροπολογία. Απλώς έχουμε τις πιο σημαντικές ομάδες τροπολογιών και τα σημεία τα οποία πρέπει να τονιστούν σε αυτό το στάδιο εξέτασης. Καταρχήν υπάρχει συμφωνία για την νομική βάση που θεωρείται δεδομένη, αλλά έχουμε συμφωνήσει για τα θέματα απάτης ΦΠΑ, που είναι οι τροπολογίες 35-38, 49 και 50. Υπάρχουν επίσης ορισμένες τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν για να αφαιρεθεί το θέμα των εσόδων που προέρχεται από την έσπαξη ΦΠΑ από την εμβέλεια αυτής της οδηγίας. Συμφωνήσαμε όλοι όμως το ΦΠΑ να περιλαμβάνεται, η απάτη ΦΠΑ να περιλαμβάνεται σε αυτό το νομοθέτημα και επίσης για το δικαίωμα των κρατών να επιβάλλουν αυστηρότερες κυρώσεις είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε μια συνενέτηση, να προβούμε σε ένα συμβιβασμό ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να υπάρχουν ευρείες εξουσίες στο εθνικό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν αυτό το κείμενο, το συμβαστικό, όπου έχει τροποποιηθεί η έννοια της αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας με την ε, ε, διατύπωση για τις υποχρεώσεις που πρέπει να δεχτούν τα κρατημέλη και η κυρία ε, Γκρέσλε έχει μια πρόταση για τις ε, ηθελημένες πράξεις δημοσίων αξιωματούχων που αφορά το σημείο 61 και υπάρχει και κάποιο περιθώριο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή συμβαστική λύση σε ό,τι αφορά την ε, ε, απαλυφή των ελάχιστων κυρώσεων και αυτό είναι ένα από τα επίμαχα σημεία γιατί εδώ μιλάμε για ποινικό δίκαιο. Είναι μια από τις πρώτες φορές που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ως νομοθέτη σε θέματα ποινικού δικαίου. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επικοινωμορφίες στα νομικά συστήματα των κρατών μελών και διαφορές, και ότι πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους και υπάρχει μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση και είναι μια ομοιόμορφη προσέγγιση για τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων και την επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά λοιπόν έχουμε αποδεχθεί την αρχή ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναφορά σε θέσπιση ελαχίστων ε, κυρώσεων σε αυτή την πρωτοβουλία. Και υπάρχει και ένα επίπεδο συμφωνίας να διαφωνήσουμε σε σχέση με το ρόλο που θα διαδραματίσει η Eurojust στο άμεσο μέλλον, αλλά και για τις τροπολογίες 96% της αναφορές που μας δίνει η Κομισιόν. Για τις τροπολογίες αυτές έχουμε καταλήξει ως συνεισηγητές σε μια συμβαστική λύση που την ανέφερε η κυρία Γκρέσλερ. Μπορώ να εκφράσω λοιπόν την ικανοποίησή μου για την συνεργασία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και των δύο επιτροπών και νομίζω και πάλι ότι έχουμε ενώπιόν μας ένα παράδειγμα που δείχνει ότι παρά την κάπως βαρία διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε λόγω των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κανονισμού μας και που πολλές φορές μπορεί να μας παγιδεύσουν, να παγιδεύσουν πάνω από μια επιτροπή σε ένα δύσκολο έργο και μας υποχρεώνουν να κάνουμε εξαντλητικές προσπάθειες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ιδιαίτερα πολυδέδαλα διαδικαστικά προβλήματα που φυσικά εμπλέκουν και θέματα ουσίας. Μετά από όλα αυτά έχουμε καταλήξει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου και συγχαίρω και ευχαριστώ όλους που ενεπλάξαν. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και τους δύο συνεισηγητές. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα προκύψει μια σημαντική πολιτική συζήτηση για τα θέματα αυτά και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και να τις αξιολογήσουμε αν το επιθυμείτε θέλει κάποιος να λάβει το λόγο σχετικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα καλά τους συνεισηγητές. Δηλαδή υπάρχει συμφωνία για την αλλαγή της νομικής βάσης με χρησιμοποίηση του 83. Όχι, από την αρχή το είχαμε θεωρήσει δεδομένο αυτό από την αρχή λοιπόν είπαμε ότι θέλουμε να επιμείνουμε στο 325 ως βάση. Και για μας της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών αυτό είναι το βασικό. Θα ψηφίσουμε χωριστά βέβαια. Καλά, συμφωνήσατε λοιπόν ότι διαφωνείτε από αυτού. Και εγώ είμαι από την Επιτροπή σας Δημοσίων Ελευθεριών και νόμιζα ότι άλλο ίσχυε, τέλος πάντων. Άκουσα τους δύο συνεισηγητές να μιλούν για ελάχιστα επίπεδα κυρώσεων ή προστήμων. Ισχύει αυτό ακόμη γιατί αν ναι, τότε είναι σοβαρό πρόβλημα για τους πράσινους. Και το είπατε και στην εισαγωγή σας ότι εδώ πρόκειται για ποινικό δίκαιο και ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε θερμοθετώντας ελάχιστα πρόστιμα ή κυρώσεις. Κατάλαβα ότι υπήρξε συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα τον δεχτούμε κι εμείς. Τρίτο και τελευταίο σχόλιο. Το θέμα των απατών σε σχέση με το ΦΠΑ. Αν συμπεριληφθεί και αυτό σε αυτή την πρόταση θα σήμαινε ότι όλα όσα αφορούν τις απάτες για το ΦΠΑ θα διώκονται ενωσιακός και όχι πλέον εθνικός διότι σύμφωνα με τον νέο, τη νέα αυτή θέση του Ευρωπαίου Ισαγγελέα θα ισχύει αυτή η δικαιοδοσία. Θα ήθελα να αποσαφινιστεί αυτό για να είμαι βέβαιη ότι υπάρχει με καταπολέμηση της απάτης για το ΦΠΑ αλλά και αναλογικότητα μεταξύ του 1% στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενώ το 99% στους εθνικούς πρέπει να γίνει σεβαστή και αυτή. Αυτό να αποσαφινιστεί γιατί βλέπω πολλές τροπολογίες από συναδέλφους για το θέμα αυτό του ΦΠΑ και των απατών. Ευχαριστούμε πολύ. Μπρατκόφσκι τώρα. Ευχαριστώ. Για την οδηγία που συζητάμε θα ήθελα να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες 35, 36, 37, 46 και 50. 47 και Καταρχήν, το η νομική βάση, δηλαδή το 113, όπου λέγεται ότι τα θέματα που αφορούν το ΦΠΑ είναι αποκλειστικό θέμα του Συμβουλίου. Μια άλλη διαφορετική νομική βάση, επομένω θα παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο ακόμα και αν υπάρχει όντως σύνδεση μεταξύ απατών ΦΠΑ και ενωσιακού προϋπολογισμού, αυτό δεν θα δικαιολογούσε η οδηγία αυτή να επεκταθεί σε όλα τα θέματα, εφαρμόζεται για όλα τα θέματα ΦΠΑ σε ολόκληρη την Ένωση, πόσο μάλλον που ο τρόπος υπολογισμού είναι πάρα πολύ πολύπλοκος από την Κομισιόν και δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Συμφωνώ ότι πρέπει να, η βάση να είναι ευρεία, αλλά επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για θέμα ποινικό και ότι επομένως δεν πρόκειται μόνο για ΦΠΑ οποιαδήποτε παρανομία βλάπτει τον προπολογισμό, βλάπτει και την Ένωση. Αλλά το θέμα των ψεύτικων λογαριασμών ΦΠΑ και η καταπολέμηση αυτής της απάτης δεν καταλήγει σε μεγαλύτερο κέρδος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εξάλλου το άρθρο 96 της συνθήκης καθορίζει το πεδίο εφαρμογής τέτοιων δικαιοδοσιών. Αν λοιπόν τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα ληφθούν υπόψη στην οδηγία για το ΦΠΑ υπάρχει διεύρυνση των δικαιοδοσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι αδύνατο διότι δεν έχει σχέση με την οδηγία. Δεν μπορούμε εξάλλου να πούμε ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι μέσα στο πεδίο γενικότερα το πλαίσιο των συμφερόντων της Ένωσης και του Κοινοβουλίου. Όχι, η συνθήκη τα πρεσβεύει αυτά. Η συνθήκη είναι η ίδια ο θέματοφύλαξη. Εξάλλου η οδηγία ως έχει θα μπορούσε να καταλήξει σε 16.000 περισσότερες υποθέσεις απάτης για το ΦΠΑ στα δικαστήρια. στο δικαστήριο. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την τροπολογία μου. Κάποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο από τις, και από τις δύο επιτροπές. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στην Σουέντερ από την Eurojust, από την ε, αρμόδια επιτροπή, ε, την αρμόδια υπηρεσία και έχουμε επίσης και εκπροσώπους της όλα η οποία μπορεί να θέλει να λάβει το λόγο. Ποιος θέλει να λάβει πρώτος το λόγο, κυρία Σουέντερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εισηγητές αλλά και τα άλλα διακεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει για να βελτιώσουν αυτή τη σημαντική πρόταση προστασίας των, συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μακρύς ο δρόμος, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Άκουσα με προσοχή τις ε, παρατηρήσεις των δύο εισηγητών και από την πλευρά της Κομισιόν μπορώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα και ιδίως και το γεγονός ότι βρέθηκε κάποια συμβιβαστική λύση για θέματα που είναι κεφαλαιόδη στην άποψη της Κομισιόν μέσα στην πρόταση αυτή. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των αδικημάτων που συνάπτονται με περιπτώσεις απάτης. Η Κομισιόν επίσης, η Επιτροπή σας μάλλον δέχτηκε να διευρύνει την εμβέλεια αυτού του νομοθετήματος που είναι κάτι πολύ θετικό για μας και δεύτερον για το καθεστώς κυρώσεων. Ξέρουμε ότι εμπλεκόμαστε φυσικά τώρα σε χώρο ποινικού δικαίου αλλά μπορούμε παρόλα αυτά να θεωρήσουμε επί τη βάση της συσσωρευμένης εμπειρίας ότι υπάρχουν κάποια αδικήματα για τα οποία χρειάζεται ένα αποτρεπτικό καθεστώς για να εμποδιστεί η απάτη. Χαίρομαι λοιπόν για τη συμφωνία των δύο συγητών για το χαμηλότερο και υψηλότερο επίπεδο κυρώσεων. Αυτό είναι φυσικά ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά αυτό το οποίο έχει παρουσιαστεί από τους συγητές είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Και φυσικά η Κομισιόν θα προσπαθήσει να διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Υπάρχει και το θέμα του χρονικού περιορισμού από ό,τι βλέπουμε από τις τροπολογίες <clears throat> κατανοούμε ότι υποστηρίζεται την Κομισιόν να υπάρχουν σαφείς κανόνες για παραγραφή αυτών των αδικημάτων που αναφέρονται στην οδηγία και αυτό είναι κατά την απόψή μας ένα από τα κύρια στοιχεία της ε, πρότασης αυτής ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα ε, υπάρχει πρόβλημα παραγραφής που θα εμποδίζει τη δίωξη αυτών των αδικημάτων. Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν, γι' αυτό χαιρόμαστε για αυτή την τροπολογία και τονίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια συζήτηση σε βάθος με το Συμβούλιο το οποίο έχει διαφορετική άποψη και πάρα πολύ σύντομα για τη νομική βάση βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν διαφορές. Η Κομισιόν παραμένει πιστή στη δική της πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 325 και θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα της νομικής βάσης αν θέλετε μπορώ να απαντήσω και το ερώτημα της κυρίας Σαρτζεντίνη για τα θέματα του ΦΠΑ και τις συνέπειες που θα προκύψουν για το μελλοντικό έργο του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Έχουμε δύο, τρόπο, δύο θέσεις. Έχουμε αυτή την πρόταση που αφορά ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και όπου λέμε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η απάτη ΦΠΑ στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια δεύτερη πρόταση για την εισαγγελική αρχή αναφέρεται με πιο εύκαμπτο τρόπο σε αυτή την οδηγία. Αυτό το οποίο όμως είναι σαφές, αν εξαιρεθεί πλήρω η απάτη ΦΠΑ από αυτήν την οδηγία, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα για να αντιμετωπίσει και να διώξει τέτοιου είδους αδικήματα που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ. Ίσως βέβαια ο οικονομικός εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να βρει κάποιες λύσεις που να λένε ότι δεν μπορεί να έχει ευθύνη η εισαγγελική αρχή για όλες τις περιπτώσεις απάντης ΦΠΑ. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από τη μορφή που θα δώσει στο, στην εισαγγελική αυτή αρχή ο Ευρωπαίος νομοθέτης με την τωρινή πρόταση της Κομισιόν θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, αυτό είναι που προτείνει η Κομισιόν όμως σε σχέση με την εισαγγελική αρχή, θα πρέπει να συζητηθεί με το Συμβούλιο καθώς και με το Κοινοβούλιο και δεν μπορώ να αποκλείσω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον. Μπορώ να φανταστώ ότι θα βρεθεί μια λύση για την πρόταση σε σχέση με την εισαγγελική αρχή που θα λέει ότι είναι υπεύθυνο για πιο σοβαρές περιπτώσεις απάτης ΦΠΑ και οι πιο ίσονες περιπτώσεις θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά αυτό και των εισαγγελικών αρχών των κρατών μελών. Αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω εάν ε, θέλει να πει κάποιος, ε, κάτι να πει κ. Σκούλα από τον ε, οργανισμό Όλαφ. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση υποστηρίζω αυτά που είπε η Αλεξάνδρα πλήρως. Να έχουμε υπόψη μας πρέπει πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια προσέγγισης ε, των νομοθεσιών στα πλαίσια ακριβώς της προσπάθειας δημιουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι αυτή η εισαγγελία θα βασιστεί στο εθνικό δίκαιο και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εθνικές εισαγγελίες σε πολλούς ε, τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα του εμπράγματου δικαίου και στις διαπραγματεύσεις ε, για το θέμα αυτό έχει υποθεί επανειλημμένα ότι η προϋπόθεση ε, για να υπάρξει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι να υπάρχει επαρκής βαθμός εναρμόνισης προσέγγισης των νομοθεσιών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό συνδέεται με όλα τα θέματα που ήδη αναφέραμε. Με βάση την ομολογία τώρα του δικαστηρίου έχει ήδη διασφαλιστεί ότι ε, ο ΦΠΑ είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του, του άρθρου 325. Και όπως είπε και η Αλεξάνδρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι προδιαγραφές του 325 παρά του 380. Το μιλάει για ουσιώδεις, αποτρεπτικές και ισοδύναμες ε, πρωτοβουλίες και μέτρα. Ενώ το 380 ε, ασχολείται μόνο με ελάχιστες προδιαγραφές. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε φιλόδοξους στόχους προσέγγισης των νομοθεσιών, τότε το 325 είναι ουσιοδός αυτονόητο. Και τονίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και πάλι η συγγήτρια, κυρία Γκρέσλε. Γκρέσλε, τι ρόλο θέλει να παίξει το Κοινοβούλιο για τη δημιουργία αυτού του δικαίου. Αυτό είναι το ερώτημα. Το 325 μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Ενώ το 380 μας αποκλείει. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πρώτα βήματα και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η Λίμπε θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο. Αυτό σημαίνει πως δεν θα επηρεάσουμε αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει λοιπόν να σας αποτρέψω πραγματικά. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Από πλευράς των συμφερόντων του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσει η Λίμπε, αλλά για μας είναι σημαντικό δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με αυτά που έχουμε ήδη. Θέλουμε οπωσδήποτε ο ΦΠΑ να συμπεριληφθεί σε αυτό το μέτρο και η σύμβαση, η συμφωνία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης λέει ακριβώς ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με το ΦΠΑ. Έχουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια διαμεθοριακής απάτης και είναι πολύ περίπλοκες οι υποθέσεις αυτές. Κανείς δεν μπορεί από μόνος του να τις παρακολουθήσει. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων μας και των κρατών μελών τα θέματα, οι ε, παραβάσεις αυτές να μπορούν να διώκονται. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια δεν θα πρέπει λοιπόν να φοβηθούμε, να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα της συναδέλφου Σαργεντίνη και καταλαβαίνω ότι θα υπήρχε κίνδυνος ε, ο Ευρωπαϊκός εισαγγελέα να αντιμετωπίζει πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα καθορίσει ο κανονισμός ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποιες αρμοδιότητες θα έχει και πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί με τις εθνικές εισαγγελικές αρχές. Θα ήθελα για το θέμα λοιπόν αυτό να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν διότι από την εμπειρία μας ε, με την Όλαφ διαπιστώσουμε, έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι είναι πρόβλημα και θα πρέπει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να τα λύσει αυτά. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ΦΠΑ από την ε, οδηγία αυτή. Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις υποθέσεις αυτές. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βεβαίως, αυτό σημαίνει επιβάρυνση, αλλά πρέπει να επιληθεί με τον κανονισμό. Οι ελάχιστε κυρώσει. Ξέρουμε για την Ολλανδία είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά πρέπει να πω ότι αν δεν προβλέψουμε μίνιμουμ κυρώσει, τότε μπορούμε να την ξεχάσουμε την υπόθεση αυτή γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο καθένα θα κάνει ό,τι γουστάρει, με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε στην εσωτερική αγορά το οργανωμένο έγκλημα θα προτιμάει τις δικαιοδοσίες που το συμφέρουν. όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να ε, διαπιστωθεί και να υπάρξουν κυρώσεις για τις περιπτώσεις απάτης. Δεν πρέπει να δημιουργούμε λοιπόν τέτοιους χώρους ε, όπου να μην ισχύει ουσιαστικά το δίκαιο στην ε, ενιαία ώρα. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό αυτό το θέμα των ελαχίστων κυρώσεων. Παρακαλώ λοιπόν. Να πω το εξή. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είπε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στην προσπάθεια διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ανεξάρτητο που να μην μπορεί κανείς να έχει τόσο ανεξάρτητη αυτή η, διαδικασία και τα άτομα που θα συμμετέχουν που να μην έχουμε καμία δυνατότητα να καταλάβουμε τι γίνεται. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ανεπαρκής. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στόχος μας πρέπει να είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Δεν μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εισαγγελία να, ε, να λειτουργεί έτσι που να είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Κατά τα άλλα, οι συμβαστικές της ΛΥΜΠΕ είναι καλές. Αλλά για το θέμα του διορισμού και το θέμα μομφής κατά ε, της Ευρωπαϊκής δεν έχουν ρυθμιστεί επαρκώς και θα ήταν δραματικό να μην εγκριθούν οι τροπολογίες μας στη ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα δύσκολο θέμα το οποίο αντιμετωπίσουμε από τη δική μου οπτική γωνία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το οποίο είπε ήδη η κυρία Σαρτζεντίνη, δηλαδή και εδώ ίσως ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ μπορεί να επανέλθει σε αυτό το θέμα, το θέμα των ελαχίστων κυρώσεων δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει οδηγήσει σε διαμάχες στις κάτω χώρες, αλλά και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν πώς βλέπει την κατάσταση στο Συμβούλιο των Υπουργών, τις συζητήσεις μεταξύ των ε, εκπροσώπων των κρατών μελών, ποια είναι η άποψή σας, γιατί εμείς φυσικά θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ορισμένοι άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η οδηγία ώστε να οικοδομηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά αυτά είναι δύο διαφορετικά εγχειρήματα. Και δεν βλέπω να υπάρχει μια σαφής και ευρία συνένεση στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Εγώ απλώς από την πλευρά των φιλελευθέρων μπορώ να σας πω ότι για μας τα θέματα αυτά είναι τελείως διαφορετικά, τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο και θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις ε, αμφιβολίες που υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Αλλά θα ήθελα να ακούσω τι πιστεύει ο κύριος Αγγιλάρ και επίσης προηγουμένως η Κομισιόν αν μπορεί να μας πει πώς εκτιμά το επίπεδο προόδου μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. κύριος Λόπες Αγγιλάρ μάλλον πρώτος. Θέλω να συνοψίσω λιγάκι τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Γκρέσλε και εγώ ως συνεισηγητές καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια γενική θέση που υπάρχουν μέσα σε αυτήν βέβαια ορισμένα σημεία που έχουμε συμφωνήσει να διαφωνούμε. Σας έχει παρουσιάσει η κυρία Γκρέσλε την συνολική προσέγγιση σε σχέση με τις τροπολογίες και εγώ αποδέχομαι την προσέγγιση αυτή σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να προσθέσω όμως ότι σε ό,τι αφορά την νομική βάση από την αρχή των συζητήσεών μας γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια σαφής ε, διαφωνία για την νομική βάση. Ξέρω ότι με τη χρήση του άρθρου 325 τα πράγματα διευκολύνονται. Πρόκειται για μια οδηγία όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ενισχυμένος. Ενώ το άρθρο 83 εμπλέκει περισσότερο <clears throat> τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί το, αυτό το εν του ποινικό δίκαιο σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά για μένα αυτή είναι η βασική ιδέα. Η ιδέα είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λειτουργήσει για πρώτη φορά ως νομοθέτης στο χώρο του ποινικού δικαίου και όχι με τρόπο ο οποίος θα είναι απεριόριστος αλλά να εστιάσει σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό θεμάτων που περιλαμβάνεται σαφώς στο άρθρο 83. Θέματα διαφθοράς, ε, τρομοκρατίας, λαθρεμπορίας ατόμων, οικονομικής απάτης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοιου είδους οικονομικά διαμεθοριακά αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 83 του Λεχθέντος όμως. Είχαμε από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου μια γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά και συμβουλές και η αρμοδιότητα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό της νομικής βάσης είναι η νομική επιτροπή η οποία είναι αρμόδια και αυτή θεωρεί ότι το άρθρο 83 θα πρέπει να είναι το άρθρο που θα χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση. Η νομική επιτροπή έχει λοιπόν αποφασίσει για το θέμα αυτό. Είναι οριστική επομένω η θέση του Κοινοβουλίου για το άρθρο 83. Γι' αυτό έχουμε παραμείνει πιστοί στο άρθρο 83. Αυτό όμως μπορεί να το διαφυσβητήσει κανείς. Δεν θα υπάρξει λοιπόν μια συνολική θέση γι' αυτό. Η κάθε επιτροπή μπορεί να κρίνει για την βάση με βάση τη δική της άποψη. Υπάρχει επίσης και μια διαφορά σε επίπεδο αποχρώσεων όταν σκεφτόμαστε για τον ενδεχόμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελικής Αρχής στο μέλλον. Για μένα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το καθήκον αυτό η εισαγγελική αρχή και να μπορέσει να υπάρξει ένα συνολικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ε, δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικού δικαίου. Να υπάρχει λοιπόν μια αρχή η οποία μπορεί να απαγγέλει κατηγορίες και να παίρνει αποφάσεις για θέματα ποινικού δικαίου τα οποία εμπλέκουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο, είναι προφανές ότι δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει κάποτε να γίνει πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ε, και επί τη βάση της ε, εμπειρία της Eurojust ως μια αρχή η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο στο μέλλον. Έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις διαφορές και έχει ληφθεί αυτό υπόψη στο τελικό σχέδιο έκθεση Σε ό,τι αφορά όμως τις απάτες ΦΠΑ και αυτό είναι το σημείο που θέλω να υπογραμμίσω, πρόκειται για έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και σε μεγάλο βαθμό πρέπει, εφόσον είναι έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της ε, οδηγίας. Οποιαδήποτε μορφή απάτηση λοιπόν ΦΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το νομοθέτημα ώστε να είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απάτη ΦΠΑ εναντίον των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έλκονται από την οδηγία αυτή που καλύπτει τα θέματα απάτη στα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισπράττει ένα ποσοστό του ΦΠΑ, το οποίο βέβαια συλλέγεται από τα κράτη-μέλη, και τα ποσά αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος για το θέμα των ελαχίστων κυρώσεων και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Αυτό είναι ο πυρήνα τη οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχουν κοινοί ορισμοί για αδικήματα, για συμπεριφορέ οι οποίε θα πρέπει να θεωρηθούν κολάσιμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγχρόνω ελάχιστε κυρώσει οι οποίες θα πρέπει αργά ή γρήγορα να ενσωματωθούν στην εθνική ε, ένωμη τάξη των κρατών μελών που δεν έχουν επιβάλει τέτοιες κυρώσεις μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η βασική μας ιδέα, αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για μια ε, δημιουργία ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου ή για νομοθεσία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ποινικά θέματα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τις ελάχιστες κυρώσει, Αυτές είναι λοιπόν οι αρχές τις οποίες θέλουμε να παραμείνουμε αμετακίνητοι και χαίρομαι για το γεγονός αυτό ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και οι δύο επιτροπές ελέγχου του προπολογισμού και δημοσίων ελευθεριών σε μια έκθεση, ένα σχέδιο έκθεση το οποίο παραμένει πιστό στην ενή αυτή. Σας ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Και τώρα η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Τόιερ για το θέμα των ελάχιστων κυρώσεων. Θέλω να τονίσω και πάλι από την πλευρά της Κομισιόν ότι υπάρχουν ε, πολλά κράτη-μέλη που έχουν τέτοιου είδους ε, κυρώσεις σε σχέση με τις απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά είναι ότι άλλα βέβαια έχουν τέτοιες πρόνοιες, άλλα κράτη-μέλη όμως δεν έχουν τίποτα τέτοιο. Και μπορεί να μην αποδεχτούν μια τέτοια αντιμετώπιση με ελάχιστες κυρώσεις. Το ερώτημα τώρα για το αν το μπορεί να υπάρξει επιβολή κυρώσεων επί τη βάση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη νομική βάση, και το 83 παράγραφος 2 και το 325 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή ελάχιστων κυρώσεων. Το 83 2 αναφέρεται σε ελάχιστες κυρώσεις και το 325 μας δίνει ευρείες δυνατότητες για να το εφαρμόσουμε αυτό σε ποινικέ διαδικασίες η κατάσταση τώρα των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών που είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστικά, για να το πω με διπλωματικό τρόπο, έναντι αυτής της πρότασης, έχουν πολλές επιφυλάξεις. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κράτη-μέλη τα οποία στρέφονται εναντίον της εφαρμογής ε, ελαχίστων κυρώσεων. Φυσικά είναι η πρώτη φορά που αποδιόμαστε σε ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά πρέπει να πω ότι το ποινικό δίκαιο είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για ορισμένα κράτη που δεν δέχονται την εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία εναντίον της πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχει ένας αριθμός κρατών που θέλουν να υποστηρίξουν τη θέση της Κομισιόν και την, απο... την θεωρούν ως ε, ορθή, αλλά βέβαια δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Τέλος, τι θα γίνει αν αυτή η πρόταση περιλαμβάνει τις ε, ελάχιστες κυρώσεις. Κατά την άποψη της Κομισιόν αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να επιβληθούν ελάχιστες κυρώσεις για οποιοδήποτε είδους αδικήματα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο αδίκημα το οποίο κολλάζεται με τον τρόπο αυτό και το να επιβληθούν ελάχιστες κυρώσεις είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αποτρεπτική δράση εναντίον αυτών των αδικημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρόκειται λοιπόν για άλλα αδικήματα, πρόκειται για ένα συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο υπάρχει αυτή η πρόταση να ε, υπάρξει κολασμός ποινικό. Και η νομοθεσία, η συνθήκη της ε, Λισαβόνας δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσει σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Ο φόβος λοιπόν μιας συλλήβδην επιβολής ποινικών κυρώσεων για όλα τα δικήματα δεν χωρεί. Εδώ από τη μέση της Επιτροπής ε, θέλει κανείς άλλο λόγο, ο κύριος Ντεγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν συγγνώμη γιατί ήρθα με λίγη καθυστέρηση. Πρέπει όμως να σας πω μερικά λόγια για τις ελάχιστες κυρώσεις. Το 12 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή μου για το ποινικό δίκαιο, για θέματα ποινικού δικαίου και η βασική ιδέα της ήταν ότι πρέπει να επιδεικνύουμε κάποια συνέπεια σε θέματα ποινικά. Συζητήσαμε τις ελάχιστες κυρώσεις για τις απάτες, για την έκθεση McIntyre δηλαδή. Έγιναν μακροσκελέστατες συζητήσεις για αυτές και τελικά η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της ΛΥΜΠΕ τάχθηκαν κατά των ελαχίστων κυρώσεων. Ένας από τους λόγους και για μένα ο σημαντικότερος ήταν ότι για να επιδειχθεί συνέπεια δεν μπορούμε να αρχίζουμε με μια πρόταση ελαχίστων κυρώσεων χωρίς να συνοδεύεται από μια οριζόντια προσέγγιση όπου να εξηγεί η Κομισιόν πώς θα εφαρμόζονται, ποια είναι τα ωφέλη και τα αρνητικά σημεία και έπειτα για ποια ακριβώς αδικήματα δικαιολογούνται και αν καταλήξουμε ότι είναι περισσότερα τα ωφέλη να εφαρμοστούν μόνο. Αυτή είναι η συνεπής προσέγγιση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η Κομισιόν ξαφνικά φέρνει δύο προτάσεις για ελάχιστες κυρώσεις για τις απάτες. Το Συμβούλιο επιμένει να μην υπάρξουν και η επόμενη πρόταση είναι τελείως διαφορετική και οι δύο συνεισηγητές του Κοινοβουλίου συμφωνούν πια για τις ελάχιστες κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι οι δύο μεγάλες ομάδες σοσιαλιστές και ΕΛΚ συμφωνούν και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ιδιαίτερα όμως για το ΕΛΚ είναι περίεργο, διότι θυμάμαι μια συνάντηση που είχαμε με την Κομισιόν για το θέμα αυτό ακριβώς. Υπήρχε μια οριζόντια ομάδα στην οποία συμμετέσχουν πολλοί και είχα ζητήσει τότε, είχα ρωτήσει, αν είναι όλοι έτοιμοι για μια οριζόντια προσέγγιση για τις ελάχιστες κυρώσεις, για τα υπέρ και τα κατά και ακριβώς το ΕΛΚ είχε ταχθεί τότε κατά. Έλεγε δεν θέλουμε ελάχιστες κυρώσεις, τελεία. Και με ιδιαίτερα που τώρα βλέπω αν και έχουν αλλάξει οι συνθήκες να βλέπω ότι ξανασυζητιούνται όλα αυτά. Ελπίζω να επιδειχθεί συνέπεια γιατί πρέπει να το ξαναδούμε. Πώς συνδέονται όλα αυτά με τις απάτες και με τη γενικότερη προσέγγιση του Κοινοβουλίου και ελπίζω τότε να μπορέσουμε να επιδείξουμε επιτέλους περισσότερη συνέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το ερώτημα, θέλει κανείς άλλο το λόγο από πλευράς των μελών της ΛΥΜΠΕ ή της ΚΟΝΤ πριν ε, να δώσω και πάλι το λόγο στους εισηγητές. Όχι. Και πάλι λοιπόν η εισηγήτρια το λόγο. να παρηγορήσω τον συνάλφο Τρέστεν. Αυτό αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι όντως κόμμα του λαού. So, Λοιπόν, δεν θα πάρω θέση, ούτε θα ζητήσω γνώμη της Κομισιόν επ' αυτού. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ο κύριος Λόπεθ Αγγελαρ για τα μέλη της ΛΥΜΠΕ στη συνεδρίαση, θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς, να φύγουμε εμείς. Εμείς, η ΛΥΜΠΕ, θα πάμε σε άλλη αίθουσα για να συζητήσουμε την, τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασής μας. Πάμε στο 4Q2, στο κτίριο Γιάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Ωραία, λίγη η κοινή συνεδρίαση. Σύντομη διακοπή. 10 η ώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού.